11 υπέρ, 30 κατά και τρεις αποχές. Και εγώ το ίδιο αποχή κράτησα. Είμαι ένας από τους τρεις. Είναι ξεκάθαρο το αποτέλεσμα, οπότε περνάμε στη ψηφοφορία της έκθεσης αυτό δεν σημαίνει, σημαίνει ότι δεν θα συνεχίσουμε το διάλογο και τις προσπάθειες. Ποιος είναι υπέρ της τροπολογίας 354. Ποιος είναι υπέρ. Υπέρ της τροπολογίας 354. Κατά. Απορρίπτεται. 46. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. Τροπολογία 491. Ποιο είναι υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Άρχεται η ψηφοφορία για την 491. Δεν σηκώσατε τα χέρια. Εγώ ξέρω να σηκώσετε τα χέρια που θα είναι το αποτέλεσμα, αλλά δεν σηκώσετε αρκετά εμφανώ τα χέρια. Τέλο ψηφοφορία. απορρίπτεται με μία ψήφο διαφορά. Συμβαστική τροπολογία 1. Άρχεται ψηφοφορία. Ηλεκτρονικά. Συμβαστική τροπολογία 1. Ηλεκτρονικά. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Περνάμε στην τροπολογία 48 τώρα. Ποιο είναι υπέρ τη τροπολογία 48? Εγκρίνεται. Η τροπολογία της Επιτροπής Περιβάλλοντος τώρα. Υπορριθμόν 29. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Περνάμε στην τροπολογία 50. Ποιος είναι υπέρ. Ποιος είναι υπέρ της 50. Εγκρίνεται. Τροπολογία 507, 508 και 509. Καταπίπτουν όμως γιατί εγκρίναμε τη 48. 51, 510, 511. Ποιος είναι υπέρ. Υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος για τις τροπολογίες αυτές. Άρχιτη ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνονται. Τροπολογία 512. Ποιος είναι υπέρ. Όχι, πάμε στην 515. Ποιος είναι υπέρ της 515. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 515. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. απορρίπτεται με τρεις ψήφους διαφορά. Τροπολογία 52. Ποιος είναι υπέρ. 52. Εγκρίνεται. Η τροπολογία 30 της Επιτροπής Περιβάλλοντος. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. 53. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. Τροπολογία 54. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 2 τώρα. Ηλεκτρονικά παρακαλώ, άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Πάμε στην 531. Δεν ψηφίζουμε για αυτήν. Οπότε πάμε στην τροπολογία 57. Ποιος είναι υπέρ της τροπολογίας 57 του εισηγητού. Εγκρίνεται. Τροπολογία έμβη, 34. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. Ελεκτρονικό έλεγχο για την τροπολογία της Επιτροπής Περιβάλλοντος. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Τροπολογία 58 του εισηγητού. Ποιο είναι υπέρ. Εγκρίνεται. Τροπολογία 59. Ποιο είναι υπέρ. Εγκρίνεται. 530 7. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. 538. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. 539. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. 541 τώρα. Ηλεκτρονικός έλεγχος προηγουμένως για την τροπολογία 539. Άρχεται η ψηφοφορία. εγκρίνεται. Στο κατάλογό σας ήταν αρχικά θετικό το πρόσημο, μετά αλλάξατε. 541 παρακαλώ, ποιος είναι υπέρ, κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος ε, για την 541, άρχεται η ψηφοφορία. Δεν ξέρω γιατί, αλλά δεν σηκώνεται το χέρι για να καταμετρήσουμε. Μάλλον εγκρίνεται, αλλά ας το ελέγξουμε. Εγκρίνεται. Τροπολογία 546. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 544 και 545. Ποιος είναι υπέρ των δύο τροπολογιών. Εγκρίνονται. 62. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. Α. Τροπολογία 63. 63. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. 64. Υπέρ. Εγκρίνεται. 65. 66 μάλλον. 66. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. 68. Ηλεκτρονικός έλεγχος πρώτα για την 66. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται. 68 τώρα. ποιο είναι υπέρ. Εγκρίνεται. 69. ποιο είναι υπέρ. Εγκρίνεται. 554. ποιο είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 71. ποιο είναι υπέρ. Εγκρίνεται. 72. ποιο είναι υπέρ. Εγκρίνεται. 73. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. 5.47 λέει ο πρόεδρος. όχι. Πάμε στην 74 κατευθείαν. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. 5.48. Ποιος είναι υπέρ. Κατά απορρίπτεται. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την τροπολογία 548. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Απορρίπτεται όπως είχε φανεί. 549. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 75. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. Τροπολογία 38 της Επιτροπής ε, Περιβάλλοντος υπέρ. Εγκρίνεται. 76. Το εισηγητό ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. Τροπολογία 550. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 77 και η 39 της ΕΜΒΗ. Ποιος είναι υπέρ εγκρίνονται. Τροπολογία 79. Ποιος είναι υπέρ? Εγκρίνεται. 557 και πανομοιότυπες. Ποιος είναι υπέρ? Αυτό είπα. 557. Ποιος είναι υπέρ? Εγκρίνονται. 57, 58, 59. 560 τροπολογία. Ποιος είναι υπέρ? κυρία Γκιλέρα λέει ότι δεν ψηφίσαμε την 532. Καλώ. το Καλώς. Ψηφίζουμε την τροπολογία 532. Ποιος είναι υπέρ. Ακαταπίπτει, καταπίπτει. Οπότε ψηφίζουμε την 560. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 560. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Και παρακαλώ και πάλι τους ε, ευρωβουλευτές Τη ομάδα μου να σηκώνουν το χέρι και ο συντονιστή του ΕΛΚ παρακαλώ να σηκώνει εμφανώ το χέρι. Πάμε στην 81. Ποιο είναι υπέρ. Εγκρίνεται. 551 και 552. Ποιο είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτονται. Τροπολογία 82. Ποιο είναι υπέρ. Εγκρίνεται. 83. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 3. Άρχεται η ψηφοφορία. Λήξη ψηφοφορίας. Εγκρίνεται, οπότε περνάμε στην τροπολογία 50 της Επιτροπής Περιβάλλοντος. Ποιος είναι υπέρ της τροπολογίας 50 της Επιτροπής Περιβάλλοντος. Κατά. Απορρίπτεται. 581 παρακαλώ. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 582. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 583. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 583. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 584. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 586. Ποιο είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 90. Ποιο είναι υπέρ. Εγκρίνεται. 587. ποιο είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 588. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 589. Ποιο είναι υπέρ. Προηγουμένω ηλεκτρονικός έλεγχος για την 588 άρχεται ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται ισοπαλία. 589 τώρα, ποιος είναι υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 91. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 590 και οι παρομοιότυπες υπέρ. Κατά. Απορρίπτονται. 52 τη Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 591. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 592. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 593. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 594 και 595. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτονται. Τροπολογία 596. Ποιος είναι υπέρ. Ε, εγκρίνεται. Οπότε πηγαίνουμε κατευθείαν στην τροπολογία 93. Ποιος είναι υπέρ. Υπέρ της 93. Εγκρίνεται. 94. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. Τροπολογία 95. Υπέρ. Εγκρίνεται. Τροπολογία 96. Υπέρ. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική τροπολογία 4. Ηλεκτρονικά άρχεται ψηφοφορία. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Και περνάμε στην τροπολογία 100. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. Τροπολογία 605. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 101. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. 102 και ισοδύναμες. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτονται. Τροπολογία 103. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. Τροπολογία 607. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 608. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 5. Άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Τέλος της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Περνάμε στην τροπολογία 618. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. Τροπολογία 619. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. 620. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 6. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Περνάμε στην τροπολογία 65. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 35. Ποιος είναι υπέρ της ΕΜΒΗ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 67. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Ελεκτρονικός έλεγχος για την 67. Άρχεται ψηφοφορία. Zamykam głosowanie. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται με μία ψήφο διαφορά. Ψηφίζουμε τη συμβαστική τροπολογία Πέντε αυτή την ψηφίσαμε μάλλον. Οπότε περνάμε στην 109 τροπολογία. Ε, 110 συγγνώμη, ποιος είναι υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 652 του κυρίου Γιάρ, ποιος είναι υπέρ, κατά, απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 7 τώρα, ηλεκτρονικά, άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται η συμβαστική τροπολογία. Οπότε περνάμε στη τροπολογία 114. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. 115 και ισοδύναμες. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνονται. Αλλά λάθος, δεν έπρεπε καν να τους ψηφίσουμε. 663. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογίες 116 και 664. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Εγκρίνονται. Ηλεκτρονικός έλεγχος για τις τροπολογίες 116 και 664. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνονται. Δεν σας τα είχα πει. Τροπολογία 665. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 666 του κυρίου Μποβέ. Ποιος είναι υπέρ? Κατά. Απορρίπτεται. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 666. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 667 και 668. Ποιος είναι υπέρ? Κατά. Απορρίπτονται. Τροπολογία 59 της Επιτροπής Περιβάλλοντος. Ποιος είναι υπέρ, κατά, απορρίπτεται. Τροπολογία 669. Ποιος είναι υπέρ, κατά, απορρίπτεται. Τροπολογία 670. Ποιος είναι υπέρ, κατά, απορρίπτεται. Τροπολογία 117 του εισηγητού. Ποιος είναι υπέρ, εγκρίνεται. Τροπολογία 117 την ψηφίσαμε. 671 παρακαλώ. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογίες. Ε, τροπολογία 674. Ποιο είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 675. ποιο είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 118. ποιο είναι υπέρ Εγκρίνεται. 676. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 119. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 677. Αλλά προηγουμένως ηλεκτρονικός έλεγχος για την 119. Άρχεται ψηφοφορία. Τέλος της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 677. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 8. Ηλεκτρονικά άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 688. Ποιος είναι υπέρ, κατά. Απορρίπτεται. 691. Α, ηλεκτρονικός έλεγχος για την 688. Θέλετε. Δεν χρειάζεται. Άντε εντάξει. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 688. Νομίζω ότι ήταν εμφανής η διαφορά. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε με διαφορά. Πάμε τώρα στην ε, τροπολογία 691. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογίες 121 και 692. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνονται. 122 το εισηγητού. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. 123 το εισηγητού. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. 124 του εισηγητού. Υπέρ. Εγκρίνεται. Τροπολογία 60 της Επιτροπής Ένδη. Ποιος είναι υπέρ, κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογίες 125 και ισοδύναμες. Ποιος είναι υπέρ, εγκρίνονται. Τροπολογία 61 της Επιτροπής Ένδη. Ποιος είναι υπέρ, κατά. Απορρίπτεται. 69 λέει ο πρόεδρος. Κατά απορρίπτεται 126 του εισηγητού ποιος είναι υπέρ εγκρίνεται 696 ποιος είναι υπέρ κατά απορρίπτεται 697 υπέρ κατά απορρίπτεται 698 υπέρ εγκρίνεται 127 του εισηγητού ποιος είναι υπέρ εγκρίνεται 128 του εισηγητού υπέρ. Εγκρίνεται. 700. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογίες 129 και 701. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνονται. Τροπολογία 130 του εισηγητού. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. 702. Ποιος είναι υπέρ εγκρίνεται. 131, 132 μάλλον και 703 υπέρ. Υπέρ εγκρίνεται. 133 ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. 134 και ισοδύναμη 704 υπέρ. Εγκρίνονται. 135 του εισηγητού ποιος είναι υπέρ Εγκρίνεται. Τροπολογία 705. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. 706 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 707 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 708. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 62 της Επιτροπής Περιβάλλοντος. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 709. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. 710. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 136 του εισηγητού. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. Τροπολογία 137. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. 138. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. 139. Πάλι το εισηγητή υπέρ. Εγκρίνεται. 140. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. 141. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. 142. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. 143 υπέρ. Εγκρίνεται. 144 υπέρ. Εγκρίνεται. 145 υπέρ. Εγκρίνεται. 146 υπέρ. Εγκρίνεται. 147. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. 716 δεν ψηφίζουμε. 148. Ποιος είναι υπέρ. 148 υπέρ. Εγκρίνεται. Εκατόν εξήντα ένα. Ποιος είναι υπέρ του συγγετού είναι, εγκρίνεται. Τροπολογία 722. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 723. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 162 του εισηγητού. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. 725. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Άλλο στο ελέγξουμε. Για καλό και για κακό. Άρχεται η ψηφοφορία της 725. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. η 725 απορρίπτεται. επανάληψη της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για την τροπολογία 725. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος της ψηφοφορίας. Οριακά απορρίπτεται. Με μία ψήφο διαφορά. Τροπολογία 163 του εισηγητού. Ποιο είναι υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 726. ποιο είναι υπέρ. Ή μάλλον Συγγνώμη, επαναλαμβάνουμε την ψηφοφορία για την 163. Άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά για την τροπολογία 163 του εισηγητού. Τέλος της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Οπότε περνάμε στη συμβαστική τροπολογία 9. Άρχεται η ηλεκτρονική ψηφοφορία για την συμβαστική τροπολογία 9. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Οπότε πάμε στην 65. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 738. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολόγια 66 της ΕΜΒΗ. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 165 το εισηγητού. Ποιο είναι υπέρ. Εγκρίνεται. 737. Ποιο είναι υπέρ. Ποιο είναι υπέρ τη 737. Κατά. Απορρίπτεται. 739. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 740. Ποιος είναι υπέρ κατά, απορρίπτεται. 741 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 742 υπέρ, εγκρίνεται. 744 και 745, ποιος είναι υπέρ, κατά, απορρίπτονται. 766, 166, ε, συγγνώμη, του εισηγητού. Τροπολογία 166 του εισηγητού υπέρ, εγκρίνεται. Τροπολογία 751 και ισοδύναμες. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Άρχεται η ψηφοφορία για την τροπολογία 751. Τέλος ψηφοφορίας. Α, με μία ψηφοδιαφορά εγκρίνεται. Γι' αυτό είπα να το ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Δεν πρόλαβα να ψηφίσω, λέει ο κύριο Άγνιου. Τα... Δεν πρόλαβα να πατήσω έγκαιρα. Προσθέστε και τη δική μου ψήφο. Yeah. Οπότε δέχομαι την πρόταση για επανάληψη της ψηφοφορία και εγώ έχω τραχιά και χοντρά δάχτυλα κύριε Άγνιο. αλλά από τα νιάτα μου. Τέλο ψηφοφορία για την 751 εγκρίνεται mm. Είπατε 651 άκουσα εγώ. Όχι, 751. Τώρα πάμε στην 753. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. 167. Ποιος είναι υπέρ. Του εισηγητού είναι η τροπολογία. Εγκρίνεται. 756. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 168. Του εισηγητού. Υπέρ. Εγκρίνεται. 757. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικά ψηφίζουμε την 757. Παρακαλώ άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 169 του το ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. 758. Ποιο είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 759. ποιο είναι υπέρ. Εγκρίνεται. Τροπολογία 68 της ΕΜΒΗ. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 170 του εισηγητού. Ποιο είναι υπέρ. Εγκρίνεται. 760. ποιο είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 761 ποιος είναι υπέρ κατά απορρίπτεται 762 ποιος είναι υπέρ κατά απορρίπτεται 171 του εισηγητού ποιος είναι υπέρ εγκρίνεται 763 ποιος είναι υπέρ κατά απορρίπτεται 764 υπέρ κατά απορρίπτεται 765 υπέρ Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 172 του εισηγητού υπέρ. Εγκρίνεται. Τροπολογία 173 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 767 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 174 του εισηγητού υπέρ. Εγκρίνεται. 175 του εισηγητού υπέρ κατά απορρίπτεται ηλεκτρονικός έλεγχος για την τροπολογία 175 Είχα συνηθίσει να γίνονται δεκτέ όλε τι τροπολογίε, κύριε Σιγητά, γι' αυτό μπερδεύτηκα. Άρχεται η ηλεκτρονική ψηφοφορία για την 175. Τέλο ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Εγκρίνεται και αυτή. Συγχαρητήρια Μα αυτό είπα και εγώ, εγκρίνεται είπα. 768. 768, ποιος είναι υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 176 και ισοδύναμες, ποιος είναι υπέρ, εγκρίνονται. Συμβαστική τροπολογία 10 τώρα, ηλεκτρονική ψηφοφορία, άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. εγκρίνεται, οπότε κάνουμε ένα άλμα στην 814. Γυρίστε σελίδα. Ποιος είναι υπέρ της 814. Ποιος είναι υπέρ της 814. Κατά. Απορρίπτεται. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 814. Παρακαλώ, άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίες Zamykam głosowanie. Τέλος Odrzucona. Πάμε στην 813. Υπέρ. Εγκρίνεται. 815. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 179 του εισηγήτου. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. 180 του το Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. 816. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 181 του το Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. 182 του το υπέρ. Εγκρίνεται. 817 και επανομοιότυπες. Ποιος είναι υπέρ, κατά, απορρίπτονται. 821. Ποιος είναι υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 820 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. Τροπολογία 73 της ΕΒΗ, υπέρ, κατά, απορρίπτεται. Τροπολογία 183 του εισηγητού υπέρ, εγκρίνεται. Τροπολογία 822 υπέρ, κατά απορρίπτεται 184 του εισηγητού υπέρ εγκρίνεται 825 υπέρ κατά απορρίπτεται 185 το εισηγητού ποιος είναι υπέρ κατά ηλεκτρονική ψηφοφορία για την τροπολογία 185 άρχεται η ψηφοφορία Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Πάμε τώρα στην τροπολογία 826. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. «828 ποιος είναι υπέρ κατά» απορρίπτεται. Τροπολογία 829. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. Έμβη 74. Αλλά προηγουμένως θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά το 829. Άρχεται η ηλεκτρονική ψηφοφορία για την τροπολογία 829. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Πάμε στην τροπολογία 74 της Επιτροπής Περιβάλλοντος. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. Τροπολογία 75 της Επιτροπής Περιβάλλοντος. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την τροπολογία 75 της Επιτροπής ΕΜΒΗ. Ποιος ε, άρχεται ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται με μία ψήφο διαφορά. 193. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 830. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 831. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 832 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 833 υπέρ. Εγκρίνεται. 834 υπέρ. Εγκρίνεται. 194 του εισηγητού υπέρ. Εγκρίνεται. 835 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 836 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 837 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 838. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 839 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 840 υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την τροπολογία 840. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται με σημαντική διαφορά και ψηφίζουμε τώρα τη συμβαστική τροπολογία 12 ηλεκτρονικά παρακαλώ άρχεται η ψηφοφορία τέλος ψηφοφορίας εγκρίνεται και περνάμε στην τροπολογία 879 μια μισή σελίδα επιδείξαμε ποιος είναι υπέρ της 879 εγκρίνεται 880 ποιος είναι υπέρ κατά εγκρίνεται 880 πρώτα όμως ηλεκτρονικός έλεγχος για την 880 άρχεται η ψηφοφορία τέλος ψηφοφορίας απορρίπτεται Τροπολογία 881. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. 205 του εισηγήτου. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. Τροπολογία 882. Ποιος είναι υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 883. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 884. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 206 του εισηγητού. Αλλά προηγουμένως θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά την 884. Άρχεται η ψηφοφορία. Άρχεται ψηφοφορία για την 884. Εγκρίνεται. Περνάμε στην τροπολογία 206. Ποιος είναι υπέρ? Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 207. Ποιος είναι υπέρ? Εγκρίνεται. 351. Όχι λάθος, λέει ο Πρόεδρος. 886. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. 208 του εισηγητού. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την τροπολογία 208. Άρχεται ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 888. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 890. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 891. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 892 υπέρ. Εγκρίνεται. 894 λέει ο πρόεδρος. Εγκρίνεται. 210 το εισηγητό. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. 211. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. 212 το εισηγητό. Υπέρ. Εγκρίνεται. Πάμε στη 213 του εισηγητού. Ποιος είναι υπέρ. Έμβιο MV82. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. 214 του εισηγητού. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. Ή μάλλον καταπίπτει. Συμβαστική τροπολογία 30. Ποιος είναι υπέρ. Άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Οπότε πάμε στην τροπολογία 216 του εισηγητού. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. Τροπολογία... Ή μάλλον πάμε στη συμβαστική τροπολογία 11. Ο κύριος Ανδρέο έχει μια προφορική τροπολογία. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ναι, ευχαριστώ Πρόεδρε. Μία προσθήκη μόνο. Πλην όμως σημαντική. Στη συμβαστική αυτή τροπολογία. Θέλω να προσθέσω το εξής. Εκεί που λέμε ότι τέτοιες ε, ειδικέ ε, συνθήκες θα εφαρμόζονται επίσης, θέλουμε να προσθέσουμε από την ημέρα της εφαρμογής του κανονισμού για τις πιο απομακρυσμένες περιοχές κτλ. Ευχαριστώ και κλείνει το μικρόφωνο του Πρόεδρου. Δεν βλέπω αντιρρήσει επί τη προφορική ε, τροπολογία, οπότε θα ψηφίσουμε τη συμβαστική τροπολογία 11 μαζί με την προφορική προσθήκη που μα έκανε ο κ. Αντρέ. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Οπότε περνάμε στην 915. Γυρίστε σελίδα παρακαλώ. Ποιος είναι υπέρ της 915. Εγκρίνεται. Πάμε στην τροπολογία της ΕΜΒΗ, την 83. Ποιος είναι υπέρ? Εγκρίνεται. ΕΜΒΗ 84. Ποιος είναι υπέρ? Κατά. Απορρίπτεται. 918 και 819. Υπέρ. Εγκρίνεται. 920. Ποιος είναι υπέρ? Κατά. Απορρίπτεται. 921. ποιο είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 220 του εισηγήτου. Ποιο είναι υπέρ. Εγκρίνεται. Τροπολογία 221 καταπίπτει. Πάμε στη 223 του εισηγητού. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. 224 επίσης του εισηγητού. Ποιο είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία. Ε, ηλεκτρονικός έλεγχος για την 224. άρχιδη ψηφοφορία. Η γραμματεία με ενημερώνει ότι δεν χρειάζεται να ψηφίσουμε το 224. Έχει καταπέσει, οπότε δεν χρειάζεται να ελέγξουμε ηλεκτρονικά το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας. Περνάμε στη 225 επίσης καταπίπτει, πάμε στη 226. 226 ποιος είναι υπέρ, εγκρίνεται. 227 ποιος είναι υπέρ, εγκρίνεται. 228 υπέρ, εγκρίνεται. 229 υπέρ. Εγκρίνεται. 230. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. 924. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 231. Του υπέρ. Εγκρίνεται. 925. 925. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικά ψηφίζουμε τι τροπολογίε 925 και 926. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλο ψηφοφορία. Απορρίπτονται. Τροπολογία 927. Ποιο είναι υπέρ. Εγκρίνεται. 932, 232, ε, συγγνώμη, λέει ο πρόεδρο. Καταπίπτει. Οπότε πάμε στην 929 Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 235 εγκρίνεται. 236 υπέρ εγκρίνεται. 237 υπέρ εγκρίνεται. 931. Ποιος είναι υπέρ. Ή μάλλον καταπίπτει, εντάξει. Πάμε στην 932 Ποιο είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 933 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 934 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 935 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 238 και 36 υπέρ εγκρίνονται. 9.38 ποιος είναι υπέρ εγκρίνεται. 9.39 ποιος είναι υπέρ εγκρίνεται. 900, 239 239 ποιος είναι υπέρ εγκρίνεται. Πάμε στη συμβαστική τροπολογία 13 άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Έχουμε προφορική τροπολογία. Παρακαλώ το συντάκτη να την παρουσιάσει. Για τη συμβαστική τροπολογία υπάρχουν 13 στο 1-4 θα θέλαμε να διαγράψουμε από την φράση μπορεί η έκθεση να συνοδεύεται έως το κομμάτι κίνδυνος επιμόλυνσης. Είναι μια συμφωνία στην οποία καταλήξαμε την προηγούμενη Τετάρτη. Δεν χρειάζεται ε, νομοθετική πρόταση. Είχαμε συμφωνήσει με τον εισηγητή. Ψηφίζουμε την συμβαστική τροπολογία 13 μαζί με την προφορική γιατί δεν υπήρχε αντίρρηση. Άρχεται η ψηφοφορία για την συμβαστική τροπολογία 13 μαζί με την προφορική. Ή μήπω υπάρχει αντίρρηση. Ο κύριος Δεκάστρο. Εμείς ε, δεν συμφωνούμε ε, με την προφορική τροπολογία επί του συμβιβασμού 13. Δηλαδή θέλουμε να παραμείνει η συμβαστική 13 ως έχει χωρίς εισαγωγή καμία τροπολογίας, τροποποίησης. Φαντάζομαι εκπροσωπείτε την ομάδα σας εδώ. Οπότε, μια και υπάρχει αντίρρηση, θα ψηφίσουμε τη συμβαστική τροπολογία 13 χωρίς την προφορική τροπολογία. Άρχεται η ψηφοφορία της συμβαστικής 13 χωρίς την προφορική τροπολογία. Τέλος. Εγκρίνεται η συμβαστική τροπολογία 13 και περνάμε στην τροπολογία 952. Ποιος είναι υπέρ? Εγκρίνεται. 954. Ποιος είναι υπέρ? Κατά. Εγκρίνεται. 955 και επανομοιότυπες. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνονται. 959. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 955 και τις ταυτόσημες. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνονται. Τώρα φάνηκε. Πάμε στην 962. 972, συγγνώμη. Τη κυρία Κέστιγκερ. 972. Ποιο είναι υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 972. Παρακαλώ, άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 973 και 974. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτονται. Τροπολόγια 242 του εισηγητού. Ποιο είναι υπέρ. Κατά. απορρίπτεται. Τροπολογία 971. Ποιο είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Πάμε στα παραρτήματα. Θα ψηφίσω μια δέσμη τροπολογιών εδώ. Ποιος είναι υπέρ. Ποιος είναι υπέρ αυτού του πρώτου μπλοκ του παραρτήματος. Εγκρίνεται. Τροπολογία της ΕΜΒΗ τώρα, 89. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. Εδώ γράφει το χαρτί μου σύντομο διάλειμμα. Να κάνουμε ένα πεντάλεπτο διάλειμμα παρακαλώ. Ε, Πρώτα όμως ε, έναν ηλεκτρονικό έλεγχο για την τροπολογία 89 της Επιτροπής Περιβάλλοντος. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλο Τέλος ψηφοφορίας. ψηφοφορία Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Πεντάλεπτη διακοπή παρακαλώ. και подъем такой Πολύ δημοκρατικά έλαβα την απόφαση για αυτό το σύντομο διάλειμμα. voit dans la croissance et la situation de la... Czas przerwy minął. Πέρασε και το διάλειμμά μας και επιστρέφουμε στη δουλειά μας. 255 λέει ο πρόεδρος του εισηγητού. Επιστρέφουμε λοιπόν, επαναλαμβάνω, και ψηφίζουμε την τροπολογία 255 του εισηγητού μαζί με την τροπολογία 88 της ΕΜΒΗ. Ποιος είναι υπέρ, κατά, απορρίπτονται. Τροπολογία 979 της κυρίας Αγγιλέρα. Ποιος είναι υπέρ, εγκρίνεται. 256 ε, του εισηγητού, ποιος είναι υπέρ, εγκρίνεται. 980 και πανομοιότυπες. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνονται. 983. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την τροπολογία 983. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 984. Ποιο είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 985 και ισοδύναμες. ποιο είναι υπέρ. Εγκρίνονται. 988 και πανομοιότυπες. Ποιο είναι υπέρ. Εγκρίνονται. 989 και 990. Ποιο είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτονται. 9.93 ποιο είναι υπέρ εγκρίνεται 9.97 έχουμε την προφορική τροπολογία εδώ του κυρίου Αντρίου. παρακαλώ έχετε το λόγο Ευχαριστώ πρόεδρε μια προσθήκη μόνο τα φυτά για πρώτες ύλες μάλλον πρώτες ύλες στηριζόμενες φυτικής προελεύσεως για ιατρικά προϊόντα κτλ. Αυτό το φυτικής προελεύσεως. Ευχαριστώ. Δεν υπάρχουν αντιρρήσεις. Οπότε ψηφίζουμε την τροπολογία με την προφορική προσθήκη. Ποιος είναι υπέρ, εγκρίνεται. Πάμε στην Τροπολογία χίλια. Ποιο είναι υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται η τροπολογία χίλια. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την τροπολογία χίλια. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται με δύο ψήφους διαφορά. Τροπολογία 1001. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 1002. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 1003. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Πάμε στη συμβαστική τροπολογία 14. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται και πάμε στην τροπολογία 1008. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. 1009. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την τροπολογία 1009. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Πάμε τώρα με δύο ψήφους διαφορά. 260 του εισηγητού. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. 261. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. 262. Υπέρ. Εγκρίνεται. 264. Υπέρ. Εγκρίνεται. 265 υπέρ. Εγκρίνεται. 266 υπέρ. Εγκρίνεται. 267 υπέρ. Εγκρίνεται. 267 λέει ο πρόεδρος, αλλά καταπίπτει είπαμε. Οπότε Και 1010 καταπίπτει. Πάμε στη συμβαστική τροπολογία 15. Άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται η συμβαστική τροπολογία 15. Και πάμε στη συμβαστική τροπολογία 16 ηλεκτρονικά άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος της Περνάμε στη 271 του εισηγητού. Ποιος είναι υπέρ παρακαλώ. 271. Κατά. Απορρίπτεται. 272 του εισηγητού υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 273 του εισηγητού υπέρ. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 272. Άρχεται η ψηφοφορία. Κατά τη γνώμη μου έχει απορριφθεί. Τέλος ψηφοφορία απορρίπτεται. 273 του εισηγητού. Ποιο είναι υπέρ. Εγκρίνεται. 274 υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 274. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Απορρίπτεται. 1033. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. 1034. Ή μάλλον 1035. 1035. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 1036 υπέρ. Εγκρίνεται. 275 το εισηγητό ποιο είναι υπέρ. Εγκρίνεται. 1037 ποιο είναι υπέρ. Εγκρίνεται. 276 το εισηγητό ποιο είναι υπέρ. Εγκρίνεται. 10.38 και 10.39. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος για τις ε, τροπολογίες 1038 και 1039. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος της ψηφοφορίας. Απορρίπτονται. Με δύο ψήφους διαφορά. Τροπολογία 277 του εισηγητού. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. 278 του εισηγητού υπέρ. Εγκρίνεται. 279 του εισηγητού υπέρ. Εγκρίνεται. 280 του εισηγητού υπέρ. Εγκρίνεται. Τροπολογίες 1040 και 1041. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτονται. Τροπολογία 281 του εισηγητού. Υπέρ. Εγκρίνεται. 282 του εισηγητού υπέρ εγκρίνεται. 283 του εισηγητού υπέρ εγκρίνεται. 284 του εισηγητού υπέρ εγκρίνεται. 1042 και 1043 ποιος είναι υπέρ Α. Λάθος καταπίπτουν. 285 285 ποιος είναι υπέρ εγκρίνεται. Οπότε πάμε συμβαστική τροπολογία 17 Άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Πάμε στην 287 του εισηγητού. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 287. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. απορρίπτεται. Τροπολογία 1050. Ποιος είναι υπέρ? Κατά. Απορρίπτεται. 1051. Ποιος είναι υπέρ? Κατά. Απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 18. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Πάμε στην τροπολογία 289 του εισηγητού. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. Πάμε στην συμβαστική τροπολογία. ή μάλλον στην τροπολογία 95 της ΕΝΔΗ. Ποιος είναι υπέρ, κατά. Τροπολογία 95 της Επιτροπής Περιβάλλοντος. Ναι, ναι, 95 ναι, της Επιτροπής Περιβάλλοντος. Ηλεκτρονικός έλεγχος παρακαλώ, η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται η τροπολογία 95 της ΕΜΒΗ. Πάμε στη συμβαστική τροπολογία 19. Άρχεται η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίες, Εγκρίνεται. Οπότε πάμε κατευθείαν στην 1069. Ποιος είναι υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 294 του εισηγητού. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Ηλεκτρονικό έλεγχο για την 294. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλο ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Τροπολογία 1070. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 1071. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. 295. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 295. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία MV 98. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 1072. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 296. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 1073. Πρώτα όμως ηλεκτρονικός έλεγχος για την 296 άρχεται η ψηφοφορία. Otwieram głosowanie nad poprawką 296. Zamykam głosowanie. Τέλος. Εγκρίνεται. Ποιος είναι υπέρ της 297 του εισηγητού. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 20. Άρχεται ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Τέλος, εγκρίνεται. Πάμε στην 1077 και τη συναφής, εγκρίνονται. 299, ποιος είναι υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 299. Άρχεται ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 1080. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. Τροπολογία 300 του εισηγητού. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. 1081. ποιο είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 21. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Περνάμε στην τροπολογία 304. Ποιος είναι υπέρ. 304 κατά απορρίπτεται. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την τροπολογία 304. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 1094. Ποιος είναι υπέρ της 1094. Ο κύριος Άγνιου. Πρέπει να ελέγξουμε, Πρόεδρε. Ζητήθηκε να ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Δεν βγήκε το αποτέλεσμα εκείνη την ώρα και μετά άλλαξε. Mm. Εγώ το παρακολουθούσα, να το δούμε την ώρα που βγαίνει. Τώρα χαίρομαι πολύ. Οκ. Okay. Okay. Przechodzimy do poprawki 1094. Ποιος είναι υπέρ, κατά. Απορρίπτεται. 1095 υπέρ, κατά. Απορρίπτεται. 1096 υπέρ. Εγκρίνεται. 1097 υπέρ κατά ηλεκτρονικός έλεγχος για την 1097 ε, άρχεται ψηφοφορία τέλος ψηφοφορίας εγκρίνεται 1099 Ποιος είναι υπέρ Κατά Απορρίπτεται 1100 και οι συναφείς ποιος είναι υπέρ κατά εγκρίνονται 305 του εισήγητο ποιος είναι υπέρ κατά εγκρίνεται 1106 ποιος είναι υπέρ ποιος είναι υπέρ της 1106 κατά Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 1106 άρχιτη ψηφοφορία. Τέλος. Απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 22. Άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά παρακαλώ. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Πάμε στην τροπολογία 105 της ΕΜΒΗ. Ποιος είναι υπέρ, κατά, απορρίπτεται. Τροπολογία 106 της υπέρ, κατά, απορρίπτεται. Τροπολογία 1110. Ποιος είναι υπέρ. Κατά, απορρίπτεται. Τροπολογία 23, συμβαστική. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά τη συμβαστική τροπολογία 23, άρχεται ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας, εγκρίνεται. Και πάμε στη συμβαστική τροπολογία 24. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. 109 της ένδυ. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 1121. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 1122 ποιο είναι υπέρ κατά απορρίπτεται έμβη 110 ποιος είναι υπέρ κατά απορρίπτεται τροπολογία συμβαστική 25 άρχεται η ψηφοφορία τέλος ψηφοφορίας εγκρίνεται συμβαστική τροπολογία 25 άρχεται η ψηφοφορία Τέλος. Έμβη 115. ποιο είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 11.40. Ε, ποιο είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 1141. Υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος για τη 1141. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Απορρίπτεται. Τροπολογία 1142. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 1146. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 1143. Ποιος είναι υπέρ. Κατά απορρίπτεται 1144 υπέρ κατά απορρίπτεται 1145. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 1145. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Πάμε στην 1148. Ποιος είναι υπέρ, κατά. Απορρίπτεται. 1149. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. Κύριε και ούτε την τροπολογία σας δεν ψηφίζετε. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Όχι, δεν χρειάζεται. Πάμε στην 118 της ΕΜΒΗ. Ποιος είναι υπέρ. Απορρίπτεται. 1151. Ποιος είναι υπέρ κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 119 της ΕΜΒΗ. Ποιος είναι υπέρ κατά. Απορρίπτεται. ΕΜΒΗ 120. Ποιος είναι υπέρ κατά. Απορρίπτεται. 1152. Ποιος είναι υπέρ κατά. Απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 26. Α, συγγνώμη. Έχουμε προφορική τροπολογία του κυρίου Ανδρέα στη συμβαστική 26. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Προτείνουμε να αποσυρθεί η πρόταση συμβιβασμού, δηλαδή ε, να ε, αφαιρέσουμε αυτή την αναφορά στα 154-115 χιλιόμετρα από την ίδια την αγρικία και μετά να αφαιρέσουμε και το τέλος της παραγράφου, στο τέλος δηλαδή μέχρι το outmost regions. Αυτή είναι η πρόταση τροπολογία. Πρόεδρε, εμείς ε, δεν συμφωνούμε με αυτή την προφορική τροπολογία. Εμείς θα θέλαμε να παραμείνει αυτή η αναφορά στην απόσταση, γιατί διαφορετικά καταρρύπτεται και όλη αυτή η ιδέα που εκφράζει η τροπολογία αυτή. Το σημείο αυτό. Musi e, sprzeciwić. Χρειαζόμαστε τρεις κατά για να μην ψηφιστεί η προφορική τροπολογία. Δεν βλέπω. Έχετε, έχετε τρεις. Ναι, υπάρχουν τρεις που είναι κατά της προφορικής τροπολογίας. Οπότε θα ψηφίσουμε τη συμβαστική τροπολογία 26 χωρίς την προφορική προσθήκη του κ. Αντρία. Ο κύριος Ταραμπέλα. Βεβαίως θα πρέπει να ε, σεβαστούμε όλους όσοι εκφράζονται κατά... Ε, εγώ ε, βεβαίως ε, είμαι σε μια περιοχή η οποία θα μπορούσε να βολευτεί ας πούμε από αυτήν την αντίθεση αλλά πιστεύω ότι αυτή η αναφορά στα 150 χιλιόμετρα Były trzy osoby przeciwne i poprawki Μα ούτω ή άλλω δεν θα μπει η προφορική τροπολογία γιατί τρει ε, συνάδελφοι τάχθηκαν κατά. Οπότε θα ψηφίσουμε αμετάβλητη τη συμβαστική τροπολογία 26 χωρί την προφορική προσθήκη. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίζουμε τέλο ψηφοφορία. Εγκρίνεται η συμβαστική τροπολογία. Πάμε στην 1158 της κυρίας Σράιερ. Ποιος είναι υπέρ της τροπολογίας 1158? Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 122. Ποιος είναι υπέρ? Κατά. Απορρίπτεται. 1159 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 1160 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 1161 υπέρ. Εγκρίνεται. 1162 υπέρ. Ή μάλλον καταπίπτει αυτή. 1163. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. MV 123. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. MV 125. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 1165. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. MV 126. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 1166. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Πάμε στη συμβαστική τροπολογία 26. Α, συγγνώμη. Έμβη 129 εγκρίνεται. 1173 ποιος είναι υπέρ εγκρίνεται. 1174 ποιος είναι υπέρ κατά απορρίπτεται 1174 ηλεκτρονικός έλεγχος άρχεται ψηφοφορία εγώ βλέπω ότι είχε απορριφθεί δεν ξέρω γιατί επιμένετε στον ηλεκτρονικό έλεγχο ορίστε απορρίπτεται πάμε στην τροπολογία 313 του εισηγητού ποιος είναι υπέρ εγκρίνεται 1175. Ποιος είναι υπέρ. Ή μάλλον λάθος. 1177 του κυρίου Γιάρ. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Λυπούμε πολύ. Πάμε Στη 1189 ποιος είναι υπέρ κατά απορρίπτεται. 1190 ποιος είναι υπέρ εγκρίνεται. 1190 ποιος είναι υπέρ απορρίπτεται μάλλον. Θέλετε έλεγχο? 133 της ΕΜΒ υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. ΕΜΒ 134 υπέρ. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 27. Ποιος είναι υπέρ να ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται. 1192. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 1193 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Έμβε 136 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 315 του εισηγητού υπέρ. Εγκρίνεται. 1194 και έμβη 137. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνονται. 1195 υπέρ κατά όχι λάθος λέει ο πρόεδρος πάμε στην 1197 του κυρίου Γιάρ ποιος είναι υπέρ της 1197 κατά απορρίπτεται 1199 ποιος είναι υπέρ κατά, απορρίπτεται. 1200, ποιος είναι υπέρ, κατά, απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 28, άσχητη ψηφοφορία. Τέλο głosowanie. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Πάμε στην 1205. Ποιος είναι υπέρ. 1205. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 1205. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλο Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Με, 26 ψήφους κατά, Πάμε στην 1206. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. 1208. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. 1209. Υπέρ. Εγκρίνεται. 1200. Ο κύριος Άγγινιου. Πρόεδρε, από περίεργεια ρωτάω. Μήπως ε, μπορούν να σηκώσουν το χέρι οι συνάδελφοι που δεν έχουν λάβει τα κείμενα των 1205 και μετά. Να το βεβαιωθούμε γιατί εγώ τουλάχιστον δεν το έχω και έχει γίνει πια ρεζιλίκη αυτή η κατάσταση. Συγγνώμη, αλλά οι συντονιστές και οι σκιώδεις δίνουν τις κατευθύνσεις για την ψηφοφορία. Αν δεν έχετε εμπιστοσύνη ούτε στους συντονιστές σας και στους σκιώδεις ηγετές, τι να πω. Νομίζω ότι του έχουμε εμπιστοσύνη γιατί εμεί του εκλέξαμε, του συντονιστέ και του και ηγητέ. Είμαι ο, ο ίδιος και δεν παρακολουθώ τον εαυτό μου, όπως βλέπετε. Όχι. Ελπίζω να μπορείτε να κατευθύνετε την ομάδα σας. Ίσως ε, να το αναθέσετε στο σκιώδη ηγητή για να κατευθύνει εκείνος ε, την ψηφοφορία των ομοειδάτων σας, ομοϊδάτων σας, γιατί είναι πιο εξοικειωμένοι και οδησηγητές και αυτοί ξέρουν πως πρέπει να ψηφίσει κάθε ομάδα. Πάμε στην τροπολογία 1200 τώρα. Ε, πάμε στην 1211, συγγνώμη, 1210 ήταν προηγουμένως, 1211 εγκρίνεται, 1212 και 1200 13 όχι καταπίπτουν. Οπότε πάμε στη 1223. Ποιος είναι υπέρ. 1223. Υπέρ κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος για τη 1223. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας, γιατί βλέπω ότι διστάζεται. Απορρίπτεται. Τροπολογία 1224 και ισοδύναμη υπέρ εγκρίνεται. Τροπολογία 1228. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Έμβη. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 318 του εισηγητού. Ποιο είναι υπέρ. Εγκρίνεται. Τροπολογία εισηγητού 319. ποιο είναι υπέρ. Εγκρίνεται. Τροπολογία 1229. Ποιο είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 1230 καταπίπτει. 1231. ποιο είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 1232. ποιο είναι υπέρ κατά απορρίπτεται 1233 υπέρ κατά απορρίπτεται 1234 υπέρ κατά απορρίπτεται 1235 υπέρ κατά απορρίπτεται τροπολογία 143 της ΕΒΗ υπέρ κατά απορρίπτεται. 1236 υπέρ, εγκρίνεται. 1237 υπέρ, εγκρίνεται. 1238 υπέρ, όχι, μάλλον 320 του εισηγητού. Ποιος είναι υπέρ της 320. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 1240. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. 1244. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 1244. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 1245 υπέρ. Εγκρίνεται. 1246 υπέρ. Okay. Which one? Okay. Three, wait, three, three, one, nine. What is? Here we go 319, 318. So we go to 1250. We go, we go to 12. Οπότε πάμε στη 1250. Ποιος είναι υπέρ? εγκρίνεται 1254 ποιος είναι υπέρ εγκρίνεται 1257 ποιος είναι υπέρ κατά απορρίπτεται 1258 ποιος είναι υπέρ κατά απορρίπτεται 1259 υπέρ κατά όχι καταπίπτει Οπότε πάμε στην 148 της ΕΜΒΗ. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 1261 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 1262 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 1263 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 1264 υπέρ. Εγκρίνεται. Έμβη 149 υπέρ. Εγκρίνεται. 1265 υπέρ. Εγκρίνεται. 1266 υπέρ. Εγκρίνεται. 1267 υπέρ. Εγκρίνεται. Πάμε στην 1270 ε, και την ε, ισοδύναμη. Ποιος είναι υπέρ, εγκρίνεται. 1272, ποιος είναι υπέρ, εγκρίνεται. 1275, ποιος είναι υπέρ, εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 29. Άρχεται ψηφοφορία παρακαλώ. Τέλος. Εγκρίνεται. Πάμε στο 322 του εισηγητού. Ποιο είναι υπέρ της τροπολογίας 322, εγκρίνεται. 323 του εισηγητού υπέρ, εγκρίνεται. 1280, ποιο είναι υπέρ, εγκρίνεται. 324 του εισηγητού υπέρ, εγκρίνεται. 150 έμβη και ταυτόσημε, ποιο είναι υπέρ, εγκρίνονται. 1283 υπέρ, κατά Απορρίπτεται. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 1283. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Οπότε πάμε στην 151 της ΕΜΒΗ. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. 1285. Ποιος είναι υπέρ και 1286 μαζί. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτονται. Έμβη 152 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 1287 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 1288 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 325 του εισηγητού υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 326 του εισηγητού υπέρ. Εγκρίνεται. 327 του εισηγητού υπέρ εγκρίνεται. 328 του εισηγητού υπέρ, εγκρίνεται. 329 του εισηγητού υπέρ, εγκρίνεται. 153 της έμβη υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 330 του εισηγητού υπέρ, εγκρίνεται. 331 του εισηγητού υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 1289 δεν χρειάζεται ηλεκτρονικό έλεγχος, αλλά αν επιμένετε, ηλεκτρονικός έλεγχος για την τροπολογία 331 του εισηγητού. Άρχεται η ψηφοφορία. Τι άλλαξαν γνώμη ελιστέ, φαίνεται. Τέλος η ψηφοφορία απορρίπτεται. Τροπολογία 1289. Ποιο είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Έμβη 154 υπέρ κατά απορρίπτεται. 1290 υπέρ κατά απορρίπτεται. Έμβη 155 υπέρ κατά απορρίπτεται. 1291 υπέρ κατά απορρίπτεται. Έμβη 156 υπέρ κατά απορρίπτεται. Έμβη δεύτερο παράρτημα ποιος είναι υπέρ κατά απορρίπτεται. Τροπολογία 332 του εισηγητού υπέρ. Εγκρίνεται. 1292 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 333 του εισηγητού υπέρ. Εγκρίνεται. 1293. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. 334 του εισηγητού υπέρ. Εγκρίνεται. 335 του εισηγητού υπέρ. Εγκρίνεται. 1296 υπέρ. Εγκρίνεται. 1297. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. 338 του εισηγητού υπέρ. Εγκρίνεται. 339 του εισηγητού υπέρ. Εγκρίνεται. 1298 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 1299 υπέρ Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 1298. Άρχεται η ψηφοφορία. 1298. 1298 άρχεται η ψηφοφορία. Για μου nie dlaczego chcemy sprawdzić. Dziękuję. Εγώ θεωρώ ότι δεν χρειαζόταν καν, αλλά εν πάση περιπτώσει, τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 1299. ποιο είναι υπέρ. Εγκρίνεται. 340 του εισηγητού υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 341 του εισηγητού υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Ένδυ 158 και ισοδύναμες. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνονται. 1302. Ποιος είναι υπέρ κατά απορρίπτεται 342 του εισηγητού υπέρ εγκρίνεται 343 του εισηγητού υπέρ κατά απορρίπτεται 1303 υπέρ κατά απορρίπτεται 344 του εισηγητού υπέρ κατά απορρίπτεται 1304 ποιος είναι υπέρ Εγκρίνεται. 13.06 υπέρ. Α, όχι, 13.07. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. 345 του εισηγητού υπέρ. Εγκρίνεται. 1308. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. 1309. Ποιος είναι υπέρ. Όχι. 1313, του κυρίου Ανδρίου και Ντενανό. Ποιος είναι υπέρ. Κατά τη 1313 μάλλον εγκρίνεται. Πάμε στην 1314. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 1315 υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος, αν και μάλλον έχει απορριφθεί, άρχεται η ψηφοφορία για την 1315. Τέλος. Απορρίπτεται. 346 του εισηγητού υπέρ. Εγκρίνεται. 1316 υπέρ κατά απορρίπτεται 1317 υπέρ κατά απορρίπτεται 1318 υπέρ κατά απορρίπτεται 1319 υπέρ εγκρίνεται 347 συγγνώμη του εισηγητού ποιος είναι υπέρ εγκρίνεται 347 Η 348 καταπίπτει. Πάμε στην, Πάμε στην 350 του εισηγητού. Ποιος είναι υπέρ της 350. Εγκρίνεται. 352 του εισηγητού υπέρ Υπάρχει πρόβλημα. Τροπολογία 352 του εισηγήτου ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. 353 του εισηγήτου ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. Τώρα, αιτιολογικές σκέψεις. Τροπολογία 355. Ποιος είναι υπέρ. Κατά απορρίπτεται. 3.56 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 3.57 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 3.58 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 3.59 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. Τροπολογία 1 του εισηγητού. Ποιο είναι υπέρ. Εγκρίνεται. 360. Ποιο είναι υπέρ. Εγκρίνεται. 361. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. 362 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 2 του εισηγητού. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. Τροπολογία 1 της Επιτροπής Περιβάλλοντος. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την τροπολογία 1 της Επιτροπής ΕΜΒΗ. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται με ισοπαλία. Τροπολογία 3 του εισηγητού. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. 364. Ποιος είναι υπέρ. Ή μάλλον 366. 366. Ποιος είναι υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 367 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. Έμβη 2. Ποιος είναι υπέρ, εγκρίνεται. Τροπολογία 4 του εισηγητού. Υπέρ, εγκρίνεται. Πάμε στην τροπολογία 6 του εισηγητού. Ποιος είναι υπέρ, Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την τροπολογία 6. ψηφοφορία. Zamykam głosowanie. Τέλος ψηφοφορίας. Przyjęta. Εγκρίνεται. Πάμε στην 373. Ποιος είναι υπέρ? Εγκρίνεται. 374 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 3.75 υπέρ. Εγκρίνεται. Α, όχι, συγγνώμη. Καταπίπτει. Οπότε πάμε στην τροπολογία 9 του εισηγητού. Ε, 3.89. Ποιος είναι υπέρ του κυρίου Λαβία. Εγκρίνεται. 12 του εισηγητού. Ποιος είναι υπέρ, εγκρίνεται. Πάμε τώρα στην 391. Μπούντα και Ταντσίλα. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. 393 υπέρ. Εγκρίνεται. 394 και MV8 υπέρ εγκρίνονται. MV9 υπέρ κατά απορρίπτεται. Τροπολογία 10 της MV υπέρ κατά εγκρίνεται. MV11 υπέρ εγκρίνεται. MV12 υπέρ κατά απορρίπτεται. 396. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 395. Ε, 37, συγγνώμη. 397. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. Όχι, λάθος. Διορθώνει η γραμματεία. Καταπίπτει. Έμβη 13. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. 3 98. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. 399 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Πάμε τώρα στην τροπολογία 17 του εισηγητού. Αλλά δεν χρειάζεται να το ψηφίσουμε. Πάμε στην 411 του κυρίου Καπούτο. Ποιος είναι υπέρ, κατά απορρίπτεται. 412 υπέρ, εγκρίνεται. Έμβη 15 υπέρ, εγκρίνεται. Τροπολογία 18 του εισήγητου υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την τροπολογία 18 του εισηγητού. Άρχεται ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 414. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 416. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 417. Υπέρ. Εγκρίνεται. 418. Υπέρ. Εγκρίνεται. 419. Υπέρ. Κατά απορρίπτεται. 420 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 421 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. Τροπολογία 20 του εισηγήτου υπέρ, εγκρίνεται. 422 εγκρίνεται. 426 ποιος είναι υπέρ, κατά, Ηλεκτρονικός έλεγχος για την τροπολογία 426. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Απορρίπτεται. Τροπολογία 427. το κυρίου Ταραμπέλα υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. «430» ή όχι καταπίπτει. Οπότε MV16 ποιος είναι ή μάλλον πρώτα η τροπολογία 24 του εισηγητού. Ποιος είναι υπέρ της 24. Εγκρίνεται. MV16 υπέρ. Εγκρίνεται και αυτή. Τροπολογία 432 Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. Τροπολογία 434. 434. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 444. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 445 του κ. Καπούτου υπέρ. 447. Μπούντα Νταντσίλα. Ποιο είναι υπέρ. Εγκρίνεται. 448 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 449 υπέρ. Κατά απορρίπτεται 4.51 υπέρ κατά απορρίπτεται MV19 υπέρ κατά απορρίπτεται 4.52 υπέρ κατά απορρίπτεται 4.53 υπέρ κατά απορρίπτεται τροπολογία 30 ε, συγγνώμη 4.54 υπέρ κατά απορρίπτεται 4.55 υπέρ κατά απορρίπτεται. Τροπολογία 33. Ποιος είναι υπέρ του εισηγητού. Υπέρ. Εγκρίνεται. 4.62 υπέρ. Εγκρίνεται. 4.63 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 4.64 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 4.65 υπέρ. Κατά. Καταπίπτει, καταπίπτει. Πάμε στην 470. Το 470 ποιος είναι υπέρ. 470 υπέρ. Κατά απορρίπτεται. Έμβη. 22 υπέρ. Εγκρίνεται. 471 υπέρ. Κατά Απορρίπτεται. Πάμε στο 379. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 40 και 480 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 481 υπέρ. Εγκρίνεται. 42 του εισηγητού υπέρ. Κατά. Άρχεται η ψηφοφορία για την τροπολογία 42. Τέλος. Απορρίπτεται. 482. Ποιος είναι υπέρ κατά. Απορρίπτεται. Έμβη 23 υπέρ. Εγκρίνεται. Έμβη 24 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 483 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 484 υπέρ. Εγκρίνεται. Στροπολογή 43 του συγκεκριτού υπέρ. Ή μάλλον δεν χρειάζεται. Πάμε στην 25 της έμβη υπέρ εγκρίνεται. Τροπολογία 26 της ΕΜΒ υπέρ, εγκρίνεται. «490. Ποιο είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 27 της ΕΜΒΗ. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Και φτάσαμε στην ψηφοφορία της νομοθετικής πρότασης όπως έχει τροποποιηθεί. Με ονομαστική κλίση παρακαλώ. Άρχεται η ψηφοφορία. Otwieram głosowanie. ψηφοφορίας. Εγκρίνεται και το σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος, πάλι με ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται. Και τώρα την απόφαση για την έναρξη των διαπραγματεύσεων με το Συμβούλιο με βάση το άρθρο 73 παράγραφος 2. Και για τη σύνθεση της διαπραγματευτικής ομάδας επικεφαλής θα είναι ο εισηγητής. Ποιος είναι υπέρ ή μάλλον ηλεκτρονικά γίνεται η ψηφοφορία, άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται και αυτή η πρόταση. Κύριε Χόισλινγκ, Έχετε το λόγο παρακαλώ. Συγγνώμη, έχουμε, έχουμε και αλλε ψηφοφορίε. Σιγά σιγά. Αλλά φαντάζομαι ο κύριο Χάουσλινγκ θέλει να πει κάτι μετά την ψηφοφορία. Θέλετε το λόγο κύριε Χάουσλινγκ. Ναι, όχι, θέλω μόνο να ευχαριστήσω παρά τις ε, ενοχλήσεις που εκφράστηκαν ε, για τη συνεργασία όλου του συναδέλφους, για την ψηφοφορία και για την ευρύτατη υποστήριξη. Ευχαριστώ θερμά. Ε, Σας ευχαριστούμε κύριε Χόισλινγκ και ευχαριστούμε θερμά και τους σκιώδεις ηγητές γιατί πραγματικά ήταν αξιέπαινοι οι προσπάθειές τους, ε, άοκνοι και πολύ δύσκολοι όλη αυτή η εργασία που έγινε. Συγχαρητήρια θερμά σε όλους λοιπόν και στη γραμματεία, στους συμβούλους, στους βοηθούς και έχετε μπροστά σας δύσκολο έργο στις διαπραγματεύσεις. Οπότε θα ληφθούν υπόψη και τα σχόλια του κ. Νίκολσον, του κ. Άγγινου και άλλων Ευρωβουλευτών ώστε στο μέλλον να αποφύγουμε επανάληψη τέτοιων καταστάσεων. Όλα αυτά τα σημειώσαμε για να βελτιώσουμε τον τρόπο εργασιών μας. Έχουμε δύο ακόμη ε, ψηφοφορίες. Καταρχήν ε, το, το σημείο 7, ρήτρε διασφάλιση και μηχανισμό κατά τη καταστρατήγηση, ο οποίο προβλέπει την προσωρινή αναστολή των δοσμολογικών προτιμήσεων τη Συμφωνία Σύνδεση μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομική Ενέργεια και Δημοκρατία τη Μολδαβία. Το λόγο έχει συντάκτηρη τη γνωμοδότηση, η κυρία Νταντσίλα. Σα ευχαριστώ πολύ πρόεδρε. Δεν είχαμε την έκθεση καιρό. Θα να ευχαριστώ του ε, συντάκτε, ε, του σκιώδη ηγητέ για τη συνεργασία του. Ευχαριστώ θερμά. Σα ευχαριστούμε. Η αρμόδια κατοσία επιτροπή είναι η Επιτροπή Διεθνού Εμπορίου. Ψηφίζουμε τη συνταγματοδότηση υπέρ. Όχι, ηλεκτρονικά πρέπει να ψηφίσουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Ηλεκτρονικά. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται η γνωμοδότηση και συγχαρητήρια κυρία Νταντσίλα. ίδια γνωμοδότηση για τη Συμφωνία Σύνδεση με τη Γεωργία για την προσωρινή αναστολή των δεσμολογικών προτιμήσεων. Εδώ η συγκεκριτής μας είναι ο κύριος Νέκοφ. Θέλετε το λόγο, κύριε Νέκοφ. Πιστεύω ότι πλέον η θέση μας είναι σαφής δεν υπάρχουν προβλήματα, δεν υπάρχουν τροπολογίες οι οποίες να είναι αμφιλεγόμενες. Υπάρχει μόνο μία τροπολογία. Ε, δεν πιστεύω όμως ότι είναι ιδιαίτερα ε, ε, σχετική. Πιστεύω ότι η πρόταση της Κομισιόν είναι καλή και θα τη στηρίξουμε. Καλώ ψηφίζουμε την τροπολογία Πόλτσακ. Ποιο είναι υπέρ. Τροπολογία 1, τον κύριο Πόλτσακ. Κατά. Εγκρίνεται η τροπολογία απόλυτα και τώρα ψηφίζουμε το σύνολο της γνωμοδότησης με την τροπολογία. Άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά παρακαλώ για το σχέδιο γνωμοδότησης όπως έχει τροποποιηθεί. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια κύριε Νέκοφ. Και ολοκληρώσαμε τις ψηφοφορίες θα περάσουμε στη συνεδρίαση των συντονιστών. Οι υπόλοιποι ραντεβού στις 3. Νομίζω ότι κερδίσατε με τον ιδρώτα του προσώπου σας ε, αυτό το διάλειμμα, την ανάπαυση. Και ευχαριστώ για τη βοήθεια και την ε, ιόβη υπομονή που δείξατε και την κατανόηση για τις ψηφοφορίες.